που είχαν την αρμοδιότητα και σύνταξη γνωμοδοτήσεων εκ μέρου των λοιπόν συναρμόδιων επιτροπών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να του ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το θέμα αυτό τη ημερησία διάταξη. και αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην συνεδρίαση, για την πειθαρχία που επιδείξατε και για την... Ε, αυτοθυσία ως προς την ε, ε, παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξάγεται ε, τώρα ή σε λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ τους Ερμηνείς,